Τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση της κυρίας Χιούμπνερ σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Πρώτος ομιλητής είναι η συγγήτρια κυρία Χιούμπνερ. Έχετε το λόγο. Thank uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι σύμφωνα με τον κανόνα 140 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να συνυπογράψει την Οργανική Συμφωνία μετά από την, την ε, διάσκεψη και τη διαβούλευση της ε, Αρμόδιας Επιτροπής της Συνταγματικής ε, και μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σήμερα έχω την τιμή να συστήνω την σύναψη της Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας ανάμεσα ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ισχύουσα συμφωνία ισχύει από το 2003. Είχαμε ακόμα την Ένωση των 15 κρατών μελών και ε, αυτό ε, ισχύει πριν από την έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Το Κοινοβούλιο επανελειμμένο συζήτησε την, διαπραγμα... τη νέα διαπραγμάτευση τη Διοργανική Συμφωνία ώστε να ληφθεί υπόψη το νέο νομοθετικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε από τη συνθήκη τη Λισαβόνα ώστε να παγιωθούν οι καλύτερε πρακτικέ αλλά και να ενημερωθεί η συμφωνία αυτή με βάση την σύγχρονη αντίληψη περιβελτίωσης της νομοθεσίας. Τον Ιανουάριο του 2015 η τότε νεοεκλεγής Επιτροπή Juncker δεσμεύθηκε να υποβάλει πρόταση για μια νέα διοργανική συμφωνία ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα, Ευρωκοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ε, συνέφερε στην ε, σχηματισμό της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις για την ε, αναθεώρηση της Συμφωνίας του 2003 τον Απρίλιο του 2015. Η σύσκεψη του Προέδρου ενέκρινε αυτή την πρόταση με αρχηγό των διαπραγματεύσεων τον Κίφερ Χόφστατ από πλευρά του Κοινοβουλίου που διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις σε στενή συνεργασία με την Νομική Επιτροπή και την Συνταγματική Επιτροπή και επίσης με τις σύσκεψη των Προέδρων. Τέλος, το Δεκέμβριο η διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε τη νέα ε, συμφωνία και την σύναψη της ε, συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας που εγκρίθηκε και από τη Συνταγματική Επιτροπή ε, και θα ψηφιστεί αύριο. Συμπεριλαμβάνει την, μια γενική εκτίμηση του αποτελέσματος και ζητεί τον αναγνώριση των, του αντικτύπου της νέας αυτής συμφωνίας, την ε, ε, <clears throat> διαθεσμική συμφωνία και Επίση, στι διάφορε νομοθετικέ ρυθμίσει. Εντοπίζει επίση διάφορα ζητήματα που θα πρέπει να αναλυθούν σε τεχνικό ή πολιτικό επίπεδο. Συστήνει την έγκριση τη συμφωνία, και περιλαμβάνει και μια εντολή ώστε η ΑΦΚΟ να εξετάσει το βαθμό στον οποίο οι τροπολογίε η ερμηνεία του κανονισμού είναι απαραίτητε για την εφαρμογή τη συμφωνία. Θα ήθελα να σα αναφέρω μόνο κάποια στοιχεία ιδιαίτερη σημασία για το Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με το περιεχόμενο τη νέα συμφωνία τις προγραμματισμός, ο τρόπος με τον οποίο η Κομισιόν θα δίνει συνέχεια στις νομοθετικές πρωτοβουλίες και αιτήματα του Ευρωκοινοβουλίου και θα δίνει διαβουλεύσεις όσον αφορά την απόσυρση νομοθετικών προτάσεων. Υπάρχουν επίσης εργαλεία για την καλύτερη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων της, διαδικασίας, της διαφανούς διαδικασίας. Έχουμε επίσης το θέμα της έκθεσης αντικτύπου, της αξιολόγησης αντικτύπου που θα πρέπει να είναι ισορροπημένη και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το κόστος της μη ύπαρξης νομοθεσίας. Ανεξάρτητη επίσης, ε, ε, επίσης θα πρέπει να γίνεται και η αξιολόγηση δικτύπου θα πρέπει να αντικαθιστά βέβαια την λήψη πολιτικών αποφάσεων. Ε, εξίσου σημαντικό είναι αυτό στο θέμα της αποφυγής της υπερβολικής νομοθεσίας, της αποφυγής υπερβολικού διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως. Σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση ή τις εφαρμοστικέ πράξεις, έχουμε προχωρήσει, αλλά το Κοινοβούλιο περιμένει γρήγορα συμφωνία ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα για τα κατάλληλα κριτήρια για τον καθορισμό εφαρμοστικών ή κατεξουσιοδότηση πράξεων ε, που θα αντιστοιχούν στο νομικό πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Κλείνω λέγοντας ότι έχοντας εξετάσει το περιεχόμενο της νέας διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή ΑΦΚΟ έχει εντοπίσει διάφορα ζητήματα που χρειάζεται να παρακολουθηθούν. Θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ανάλυση σε μια έκθεση κοινή πρωτοβουλία μεταξύ των ε, επιτροπών νομικών υποθέσεων και συνταγματικών υποθέσεων. Πιστεύουμε ωστόσο ότι αυτή η διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας θα είναι ένα σημαντικό μέσο για τη βελτίωση των σχέσεων και της διαφάνειας ανάμεσα στα θεσμικά όργανα ώστε να βελτιωθεί η νομοθεσία προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Και τώρα λόγος στον Υπουργό, την Υπουργό Χένης ε, Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που ξαναβρίσκομαι σε αυτή την Ολομέλεια, την ολομέλεια. Κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, η διαθεσμική συμφωνία είναι ένα λόγο για τον οποίο εμεί οι νομοθέτε ε, συναντηθήκαμε και επιβεβαιώσαμε την διάθεση συνεργασία μα. Είναι ένα σημαντικό βήμα πρόοδου στι διαθεσμικέ μα σχέσει. Με αυτή τη νέα συμφωνία από κοινού έχουμε καθορίσει ένα σύνολο κανόνων για το πώς να πετύχουμε αποτελέσματα για τους πολίτες μας και τα συμφέροντά τους. Από κοινού δεν θα επαναλάβω τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, απλώς κάποιες παρατηρήσεις για να το αποδείξω. Θα έχουμε μια κοινή συζήτηση για τις νομοθετικές μας προτεραιότητες και θα επιλέξουμε αυτές που βάσει των απόψεων των τριών θεσμικών οργάνων θα πρέπει να είναι οι κατεξοχήν προτεραιότητες για τα επόμενα τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κάποιες φορές περιγράφεται ως κατακαιρματισμένη. Πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε εδώ ενότητα και να αποστέλουμε ένα μήνυμα πυγμής ε, αντιμετωπίζοντα τις προκλήσεις που ε, παρουσιάζονται μπροστά μας με τρόπο κοινό, ενιαίο. Ω προ τι μελέτε αντικτύπου, συμφωνήσαμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να βασίζεται σε αποφάσει με τα Οπότε πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι οι διαδικασίε αυτέ είναι πολιτικού χαρακτήρα και όχι τεχνοκρατικέ. Ω συνομοθετέ έχουμε ευθύνη και καθήκον προ του πολίτε μα να διασφαλίσουμε ότι όταν λαμβάνουμε αποφάσει έχουμε διαθέσιμε όλε τι απαραίτητε πληροφορίε και ότι λαμβάνουμε υπόψη τα στοιχεία που μελετούμε. Γι' αυτό έχουμε δώσει σωστά έμφαση στο να δίνεται έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς είναι καθοριστική σημασία για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Έχουμε δεσμευτεί να αποφύγουμε την υπέρμετρη ρύθμιση και το υπέρμετρο διοικητικό άκτο. Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις καλές επιδόσεις είναι στα πλαίσια ακριβώς αυτής της συμφωνίας. Ο κατάλογο προτεραιοτήτων μα δεν πρέπει να γίνει αντιληπτό ω προσπάθεια υποβάθμιση των προτύπων αλλά το αντίθετο, θα πρέπει να σκεφτόμαστε δύο φορέ και να είμαστε προσεκτικοί ε, πριν ε, προβλέψουμε νέα νομοθεσία, εφόσον είναι απαραίτητη, για το κατά πόσο είναι απαραίτητη ή όχι. Πάντως, ε, μπορέσαμε και τι προτεραιότητε του Κοινοβουλίου να τι ενσωματώσουμε στη συμφωνία, επικεντρωνόμενοι στη σωστή μέθοδο. Θα είναι μια κοινή πλατφόρμα αυτή τη συμφωνία για τη συζήτηση για το πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε καλύτερα ότι έχουμε νομοθεσία που εξυπηρετεί τον επιδιωκόμενο σκοπό, χωρί περιττό άχθος ε, εις βάρο των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων δικήσεων. Επίσης, συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τη διαφάνεια του έργου μα για του πολίτε. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να τονίσω ότι θα έχουμε μια κοινή βάση δεδομένων για την κατάσταση των πραγμάτων ως προς τις νομοθετικές εξελίξεις. Αυτό μπορεί να ακούγεται ως ένα θέμα γραφειοκρατικό για κάποιους από εσάς. Όμω είναι σημαντικό. Οι πολίτε πρέπει να μπορούν να κατανοήσουν πώ εργαζόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαστε πιο δραστήριοι με κοινέ προσπάθειε επικοινωνία. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Το Κοινοβούλιο έχει συμφωνήσει σε πολλά σημεία μαζί μα, όπου και εμεί ω νομοθέτε θέλουμε να ενδυναμώσουμε την συνεργασία μα. Όπω το να είμαστε καλύτεροι και να δοθούμε ότι υπάρχουν αποτελεσματικότερε διαδικασίε, διασφαλίζοντα την ποιότητα τη νομοθεσία και σεβόμενοι τις, τα προνόμια και τι αρμοδιότητε ε, του καθεθεσμικού οργάνου. Γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε τη συνεργασία σε αρχικά στάδια για να καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι απόψει και τι τοποθετήσει των ΜΕΝ και ΔΕ και να διευκολύνουμε τι διαπραγματεύσει. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να εκφράσω την ε, εκτίμησή μου για την επικοδομητική στάση και του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να καθορίσουμε μέτρα και να προβλέψουμε να ε, έχουμε μάλλον περισσότερη εμπιστοσύνη σε επίπεδο κατώμελων με τι κατεξουσιοδότηση πράξη. Πρόεδρε, είμαι πεπισμένη ότι η συμφωνία αυτή θα συνεισφέρει στο να έχουμε ένα πλαίσιο και μια ατμόσφαιρα που θα ευνοήσουν τι διαπραγματεύσει και θα επιτρέψουν να έχουμε επικοδομητικότερε αποτελεσματικέ λύσει στα κοινά μα προβλήματα. Ναι, Όλοι γνωρίζουμε ότι η συμφωνία είναι αποτέλεσμα συμβιβασμών, όχι ε, κάτι που μπορεί να ικανοποιεί πλήρω τι επιμέρου ε, προτεραιότητε του κάθε θεσμικού οργάνου. Κάποια σημεία ήταν δύσκολα, ε, ευαίσθητα, λόγω τη εξισορρόπηση δυνάμεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Πιστεύω, ωστόσο, ότι η συμφωνία αντικατοπτρίζει μια δίκαιη ισορροπία. Και η θέση του Συμβουλίου για τη συμφωνία στι 15 Μαρτίου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα εγκριθεί επισήμω. Μετά θα πρέπει να περάσουμε γρήγορα στην υλοποίηση, ώστε ο ρυθμός που έχουμε ήδη αποκτήσει και εκτεμένη ταχύτητα να ε, αξιοποιηθεί για να ωφελήσουμε με την υλοποίηση των στόχων μας τους πολίτες και τις ε, επιχειρήσεις. Η ε, παρακολούθηση της υλοποίησης θα είναι μια από τις πρώτες προτεραιότητες του Συμβουλίου και την επόμενη εβδομάδα θα αποφασίσουμε πώς θα διοργανώσουμε τον τρόπο που θα εργαστούμε με βάση το πρόγραμμα εργασίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για να ανοίξουν και τριμερείς συζητήσεις για τις αιτήσεις κοινέ μας προτεραιότητες. Είμαστε στα πρώτα στάδια τη συζήτηση στο Συμβούλιο για την υλοποίηση. Ωστόσο, η Προεδρία όλο ιδιαίτερο σκοπεύει να δει πώ το Συμβούλιο θα ασχοληθεί με τι μελέτε αντικτύπου στο μέλλον και πώ θα προωθήσει το πακέτο για την καλύτερη νομοθεσία όπω έχει υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, η Προεδρία την διαφάνεια θα την φέρει μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων. Ολοκληρώνοντα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θυμίσω ότι η Προεδρία του Συμβουλίου βεβαίω θα συνεχίσει να συνεργάζεται ε, στενά με το Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βεβαιωθεί ότι υπάρχει πραγματική και ουσιαστική υλοποίηση αυτή τη τόσο σημαντική συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγο στον Επίτροπο Τίμερμαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όταν καλύτερα το σε συμφωνία το Δεκέμβριο, υπήρξαν δύο γνώμες. Εγώ χαιρόμουν που είχαμε αυτή τη συμφωνία που μας προχωρούσε αρκετά βήματα. Προσωπικά όμως θα ήθελα μια πιο φιλόδοξη συμφωνία σε πολλούς τομείς. Επικράτησε όμως ο ρεαλισμός. Ήταν και αδύνατο να πείσω τους άλλους να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο και έτσι δεχθήκαμε μια συμφωνία καλύτερη πάντως από αυτή που είχαμε πριν. Για μένα παραμένει μισογεμάτο το ποτήρι. Γιατί είναι σημαντικό λοιπόν. Γιατί πρέπει να κοιτάξουμε την, τον όλο κύκλο πολιτικής. Πρέπει δηλαδή να επανεξετάσουμε όλα όσα πράττουμε νομοθετώντας και τα τρία θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία. Ήταν ε, ε, δυσαρεστημένα και τα τρία θεσμικά όργανα με τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι τότε διαγνώσει και επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω και να τονίσω από τις τρεις διαφορετικές προοπτικές ότι κανείς δεν ήταν 100% ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της υπραγμάτευσης. Υπογραμμίζω όμως κάποια από τα αποτελέσματα που έχουν πιστεύω ουσιαστική σημασία για τις καταξουσιοδότηση ε, πράξεις υπάρχει η ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ συνομοθετών και απεμπλοκή ορισμένων ε, φακέλων. Πρέπει η Επιτροπή να εξασφαλίσει περισσότερη διαφάνεια επιτρέποντας τους εμπλεκόμενους φορείς να εξετάζουν τις κατεξουσιοδότηση ε, πράξεις και στον πολιετή προγραμματισμό και τις εφαρμοστικές πράξεις βεβαίω. Και πρέπει να προσδιοριστούν προτεραιότητες για τον ετήσιο και πολιετή σχεδιασμό και την νομοθετική διαδικασία. Για την ρυθμιστική ευρωστία θα πρέπει να εξετάζεται η παρακολούθηση κάθε νομοθετήματος στο μέλλον ώστε να βεβαιωνόμαστε ότι λειτουργεί όπως και προγραμματιστεί. Αυτό το πρόγραμμα ευρωστίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει ουσιαστικό ρόλο και στην απλούστευση της φυσταμένης νομοθεσίας, την απίσχνασή της και την ελάφρυνση του γραφειοκρατικού βάρους χωρίς ωστόσο να υποβαθμιστούν ε, ρο, ε, στόχοι πολιτική, περιβαλλοντική και άλλη. Αυτό ήταν που μας φόβησε στην αρχή, ότι μπορούσε δηλαδή να υποβαθμιστούν τα επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος κυρίως. Επίσης, κοινέ πλατφόρμες μηχανογράφησης για τις κατεξουσιοδότηση και ίσως στη συνέχεια για την διαδικασία της συναπόφασης θα επέτρεπε να ανοίξει και στη δημόσια εξέταση στο βλέμμα του κοινού αυτή η διαδικασία συνομοθετική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνεχίζει να εφαρμόζει πλήρως δεσμεύσεις της και είναι ε, απόλυτη προσήλωση της Επιτροπής σε αυτόν τον ακρογωνίο λίθο. Είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, το επαναλαμβάνω και ότι δεν ικανοποιήθηκαν όλες μου οι προσδοκίες, ισορροπημένο αποτέλεσμα προ όφελο και των τριών νομοθετικών οργάνων, ε, οργάνων που συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία και πιστεύω ότι και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να την υποστηρίξει. Ευχαριστώ την κυρία Χιούμπνερ για την εξαιρετική εκθεσή τη. Υπάρχει ένα σαφέ πολιτικό μήνυμα από τα τρία θεσμικά όργανα ότι εξετάζουμε σοβαρότητα την καλύτερη νομοθεσία, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, τον απλό άνθρωπο, γυναίκα και άντρα, είναι και 8 Μαρτίου, Θέλουμε να τον απαλλάξουμε, να την απαλλάξουμε από περί την νομοθεσία. Θέλουμε λοιπόν καλύτερη νομοθεσία από όλα τα θεσμικά όργανα ως ένα μέτρο για πιο αποτελεσματικό τρόπο ρύθμιση των διαφορών τομέων. Και αν ακολουθήσει και η συμφωνία του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να ξεκινήσει και να προχωρήσει σε συνεργασία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ταχύτατα την υλοποίηση αυτή τη πρόταση για το καλό των πολιτών και των επιχειρήσεών μα. Η Επιτροπή ιδιαίτερω μπορεί να υλοποιήσει αμέσως της δεσμεύσεις της σε σχέση με τις προτάσεις που βασίζονται στη συνθήκη της Λισαβόνας με ένα νέο μητρό κατά συμπράξεων που επίσης επιδιώκει το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Τίπερμαν για αυτή την πρωτοβουλία, ε, την πολύ σημαντική. Να συγχαρώ επίσης την κυρία Χόπνερ για την έκθεσή της που είναι δύσκολο στην ε, σύνταξή της και στην ολοκλήρωσή της. Ε, τελικά όμως είχε αίσια έκβαση και τα κατάφερε εκείνη και να συγχαρώ και τον συνάδελφο Μάρκος Πίπερ γιατί δεσμεύτηκε ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι ε, σωστά προστατευμένες στο πλαίσιο αυτής της διοργανικής συμφωνίας και τελικά να οδηγηθούμε στη νέα δεύτερη έκθεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, στη, τα αιτήματα δε του ΕΛΚ ε, εισακούστηκαν και γι' αυτό είμαστε ικανοποιημένοι. Οι αξιολογήσεις αντικτύπου είναι απαραίτητε ε, για να υπάρχει η ποιότητα και για να μην αυξηθεί ο φόρτος των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων. Θα πρέπει δηλαδή να νομοθετούμε μόνο εκεί όπου υπάρχει έλλειψη και γι' αυτό και χαίρομαι για τα όσα άκουσα από τον κύριο Τίμερμαν, γιατί είναι η κατάλληλη στιγμή για να αληθούν ε, οι δυσκολίε τι οποίε αντιμετωπίζει το Ευρωκοινοβούλιο σχεδόν σε όλε τι διαπραγματεύσει τη τελευταία δεκαετία. Και για το Ηνωμένο Βασίλειο, όντω θα πρέπει να απεφευθούν οι μη απαραίτητε νομοθεσίε, αλλά να βελτιωθεί. Και έτσι και η οικονομική ανάπτυξη είναι σημαντικό για το Ευρωκοινοβούλιο να εργαζόμαστε σε ισότιμο πεδίο. Και γι' αυτό και ακριβώ είμαστε το Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόρμπετ. Πρόεδρε, Καταρχά, θα ήθελα να καταστήσω σαφή τη θέση τη σοσιαλιστική ομάδα στη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Φυσικά είμαστε υπέρ βελτιωμένου και καλύτερου συστήματο για του νομοθέτε, ώστε να γνωρίζουν τον αντίκτυπο των όσων κάνουν και το, το πιθανό κόστος που μπορεί όλα αυτά να σημαίνουν. Βεβαίως, όμως Ανέκαθεν λέγαμε πως αυτό θα πρέπει να είναι μια συνολική αξιολόγηση. Δεν πρόκειται μόνο για την περικοπή κόστους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ε, αν και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά επίσης αφορά το κόστος και το άχθος άλλου είδους, όχι μόνο της νομοθεσίας, αλλά και το κόστος της έλλειψης νομοθεσίας. Κόστος για τον καταναλωτή, για τη δημόσια υγεία και άρα και για τον δημόσιο προϋπολογισμό, κόστος για το περιβάλλον, κόστος για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ε, πολιτική ανταγωνισμού. Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Οι αξιολογήσει αντικτύπου λοιπόν θα πρέπει να είναι καθολικές, θα πρέπει να είναι δηλαδή μια πραγματική μελέτη κόστους ωφέλειας να λαμβάνουμε επίσης το ότι νομοθετούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν κάνουμε σωστά την νομοθεσία, όταν δηλαδή ισχύουν κοινοί κανόνες για την κοινή μας αγορά, αντικαθιστούμε 28 διαφορετικές και αντιφατικές ε, εθνικές νομοθεσίες. Δηλαδή απλοποιούμε τα πράγματα για τις επιχειρήσεις, περικόπτουμε την γραφειοκρατία. Και αυτό θα πρέπει να είναι κομμάτι της εξίσωσης και η τρίτη μας ε, θέση θα πρέπει να είναι ότι θα πρέπει να είναι συμβουλευτική η άποψη της Κομισιόν. Δεν μπορεί να θέσει βέτο ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των λαών. Εμείς θα πρέπει να έχουμε την τελευταίο λόγο. Φανταστείτε πριν 30 χρόνια επειδή είναι και η Διεθνής Μέρα της Γυναίκας, ε, να λέγανε «Α, η ε, ε, μισθή για ίση εργασία, αυτό θα κοστίσει περισσότερο, άρα ας μην το κάνουμε». Και φυσικά θα έπρεπε εμείς να ξεπεράσουμε αυτή την γνώμη και να αποφασίσουμε ούτως ή άλλως. Η ομάδα μου λοιπόν, εφόσον αυτή η συμφωνία συμφωνεί για όλα αυτά και για το προγραμματισμό, τη διαφάνεια, τις αξιολογήσεις αντικτύπου και την εγκρίνουμε, και θα εργαστούμε για την περαιτέρω εφαρμογή αυτής της σημαντικής συμφωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μάκιντάιρ. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω τη συμφωνία. Πρόκειται για ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, αλλά όπως και ο Επίτροπος θα προτιμούσε να ήταν πιο φιλόδοξη. Η μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελέσει μια συνεχιζόμενη διαδικασία, δεν μπορεί να σταματήσει με αυτή τη διοργανική συμφωνία. Η περικοπή, ο περιορισμός του διοικητικού ε, κόστους επιβάρυνσης της γραφειοκρατίας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει τεράστια σημασία για την ανταγωνιστικότητά μας σε μια παγκόσμια οικονομία. Η ομάδα μου έχει καταγράψει τρεις βασικές προτεραιότητες για την διοργανική συμφωνία. Την ανταγωνιστικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το στόχο μείωσης της επιβάρυνσης και το Συμβούλιο επαλήθευση τη νομοθεσία. Εδώ στο τελευταίο σημείο προβλέπεται η θέσπιση του Συμβουλίου αυτού ως ένα ευπρόσδεκτο πρώτο βήμα για την επίτευξη της ανεξαρτησίας του. Για τους δύο πρώτους στόχους, με Συμφωνία καταγράφει τα συμπεράσματα και αντανακλά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ιδιαίτερα στον περιορισμό του βάρους. Και αυτό ήταν ένα από τα κύρια σημεία των διαπραγματεύσεων του Πρωθυπουργού της χώρας μου. Προορισμός δηλαδή του ε, στόχου και περικοπή της γραφειοκρατίας που θα είναι προς όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρης. Αυτό είχε καταστήσει σαφές ο Πρωθυπουργός της χώρας μου ότι κάνουμε την Ευρώπη καλύτερη και όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι λοιπόν η συμφωνία αυτή με την εξέταση συνεπειών, με την ρήτρα θέση εκτός λειτουργίας με μια σαφή δέσμευση υπέρ τη καταργήση των περιττών ρυθμίσεων. Με ικανοποίηση βλέπω ότι θέλει μια ετήσια επισκόπηση έκθεση επισκόπησης ε, της επιβάρυνσης από την φυστόμενη νομοθεσία έτσι ώστε και η Επιτροπή έτσι ώστε να επανεξεταστεί και η ισχύουσα νομοθεσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι σε καλύτερη θέση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι η μεταρρύθμιση έχει ζωτική σημασία. Αποτελεί μια ακόμη κίνηση προς την ορθή κατεύθυνση σε μια συνεχιζόμενη πορεία προς τη μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Φούμπνερ που είναι και πρόεδρο τη Επιτροπή, ανέφερε απόλυτα ε, σωστά ποιο είναι ο στόχο αυτή τη έκθεση που θα, θα ψηφίσουμε αύριο και εμεί θα την υπερψηφίσουμε για να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτή η διοργανική συμφωνία. το να νομοθετεί κανεί δεν είναι εύκολη δουλειά και το να νομοθετεί για 500 εκατομμύρια Ευρωπαίου σε 28 χώρε είναι ακόμα πιο δύσκολο. Πέρα από την αρχή τη ε, επικουρικότητα, τη αναλογικότητα. Ε, είναι ο στόχο μα να έχουμε νομοθετήσει νομοθεσία ποιοτική και να, μην είναι, και να είναι εύκολη στην κατανόηση και στην εφαρμογή της. Ε, αυτό σημαίνει κατανόηση των κανόνων αλλά και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους νομοθέτες, εφαρμογή και δυνατότητα εφαρμογής της νομοθεσίας που θα εγκρίνουμε, εκτίμηση των αντικτύπου και κόστος της μη ύπαρξης νομοθεσίας για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνήθως είναι ξεχασμένες στις νομοθεσίες και στις ευρωπαϊκές πολιτικές να μην επιβαρυνθούν υπέρ του θέοντος. Δεν είναι εύκολο να νομοθετεί κανείς γιατί τα γρανάζια της νομοθεσίας είναι πολύ περιπλοκά και είναι σίγουρο ότι πολλές φορές οι Ευρωπαίοι πολίτες μας βλέπουν λες και είμαστε κάπου σε κάποιο μακρινό γαλαξία κατεστημένοι. Εμείς θεωρούμε, αισθανόμαστε την ανάγκη και έχουμε συνεργαστεί στο να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ε, συμπολιτών μας με αυτή τη διοργανική συμφωνία. Νιώσαμε κάποιους από τους φραγμούς που εντοπίσαμε και διαπραγματευθήκαμε ε, ε, καλύτερη, την καλύτερη νομοθεσία. Ε, θέλουμε να υπάρχουν εξολογήσεις αντικτύπου, διαφάνεια και μείωση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων, πράγμα που θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία και καταπολέμηση της απορρίθμισης, που δεν είναι το ίδιο να νομοθετεί κανείς υπερβολικά, να νομοθετεί σωστά πρέπει κανείς, ούτε πολύ ούτε λίγο. Ωστόσο υπήρξε πίεση από πλευράς των λαϊκιστών, ενώ εγώ πιστεύω πως έχουμε καταφέρει μια ρεαλιστική ε, συμφωνία που θα προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σταθερό ε, νομοθετικό πλαίσιο. Και γι' αυτό και θα το υπερψηφίσουμε αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρυσόγονος. Συζητούμε σήμερα για τη συμφωνία μεταξύ της ευρωπαϊκής επιτροπής του ευρωπαϊκού συμβουλίου και του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου σχετικά με τη βελτίωση των εσωτερικών νομοθετικών διαδικασιών με στόχο την ορθότερη λειτουργία των οργάνων την καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών της ένωσης και την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. μετά από μακρές διαπραγματεύσεις έχουμε επιτέλους μια πρόταση με ορισμένα θετικά στοιχεία. είναι όμως φανερό πως και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οικονομικά και όχι κοινωνικά ζητήματα. οι συνδικαλιστικοί φορείς που εκφράζουν τις ανάγκες των εργαζομένων φαίνεται να τίθενται στο περιθώριο. παράλληλα γεννώνται ερωτηματικά σχετικά με το αν όντως ενισχύεται η φωνή του κοινοβουλίου κατά την νομοθετική διαδικασία ή αν αντίθετα είναι η επιτροπή εκείνη που βγαίνει κυρίως ενισχυμένη από αυτή τη συμφωνία καθώς η ευρώπη βιώνει έναν έντονο προβληματισμό για το μέλλον της θα έπρεπε να είχαμε αλλάξει στόχευση και αντιλήψεις και να εστιάσουμε στα προβλήματα των πολλών όχι στα συμφέροντα των λίγων. αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πραγματικά δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες και όχι με συμφωνίες που περιορίζουν τη φωνή των πολιτών και των οργάνων που τους εκπροσωπούν άμεσα. οι διευκολύνσεις για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την ευρωπαϊκή ένωση ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατία και να αποδυναμωθεί η γραφειοκρατία. ευχαριστώ. Επόμενος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πίσω από τα λόγια καλύτερη νομοθεσία κύριε Τίμερμανς ποιος θα μπορεί να μας πει πραγματικά εάν θα ήθελε κάποιο να νομοθετεί χειρότερα. Εγώ πιστεύω πίσω από τα λόγια αυτά κρύβεται μια ιδεολογία ολόκληρη. Η ιδεολογία της λιγότερης νομοθεσίας, όχι της καλύτερης. Αυτή που θεωρείτε και το είπατε κι εσείς, χρησιμοποίησατε τη λέξη και το έχουμε ακούσει να επαναλαμβάνετε πολλές φορές, ιδίω από τα δεξιά αυτή τη ε, ε από τη δεξιά πτέρυγα, το διοικητικό άχθο. Εγώ σα λέω, κύριε Επιτροπέ, το άχθο τη Ευρώπη δεν είναι γραφειοκρατικό. Είναι δημοκρατικό, είναι κοινωνικό, είναι τα 27 εκατομμύρια άνεργοι, είναι οι πρόσφυγε, του οποίου δεν μπορούμε να υποδεχτούμε εξωπρεπώ. Είναι τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει αυτή η Ευρώπη, που δεν έχουν κανένα γραφειοκρατικό χαρακτήρα. Πίσω λοιπόν από τις ιδεολογίες, ε, αυτό που υποκρύπτεται είναι η ιδεολογία της λιγότερης νομοθεσίας. Θέλετε να απελευθερωθεί η αγορά, ώστε η αγορά αυτή να είναι τελείως ανοιχτή. Αλλά πρέπει να ε, διαρωτηθούμε ποια Ευρώπη θέλουμε. Ευρώπη που νομοθετεί, γιατί όχι. Αυτή την Ευρώπη προασπίζομαι εγώ. Θέλουμε ποιότητα ε, στον ατμοσφαιρικό αέρα, στο νερό, τη υγεία των πολιτών που πρέπει να τη σεβόμαστε. Δεν είναι η Ευρώπη τη γραφειοκρατία που θα πληρώνουμε υπαλλήλου για να κοιτάζουμε ε, πώ δεν θα νομοθετούν για περίπου ένα χρόνο. Ο Κάφκα το είχε οραματιστεί αυτό και η Ευρώπη το πραγματοποιεί. Και τώρα η κυρία Ντινόλφη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Η συμφωνία που τώρα ετοιμαζόμαστε να εγκρίνουμε είναι αποτέλεσμα συμβαστική ε, λύση, αλλά προ τα χείρο. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με εμά ω άμεσα εκλεγμένου προσώπου των πολιτών, θα ήθελε να πετυχαίνει περισσότερα. Αυτό μα ζητάτε. Η συμβαστική λύση που επιτέχθηκε δεν είναι από τι καλύτερε. Εμεί ω κίνημα πέντε αστέρε θα ζητούσαμε λόγω χάρη περισσότερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά του τριμερεί διαλόγου. Δεν ε, αρκεί να ξέρουμε τι αποφασίστηκε εκ των υστέρων. Οι πολίτε πρέπει να γνωρίζουν τι είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση από την αρχή. Επίση, μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών τα ειδικά μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά, η μεγαλύτερη προβολή και διαφάνεια για τις κατακρισοδότηση και εφαρμοτιστικές πράξεις. Ε, επίσης να μην προκύπτουμε μόνο στις πιέσεις των ε, ομάδων των λόμπι γιατί αυτό φαίνεται ότι πιο πολύ μας επηρεάζει επίσης για την κατεξουσιοδότηση πράξης δεν καταλαβαίνουμε γιατί ε, όλες αυτές οι ρυθμίσεις θα αρχίσουν να ισχύουν μόλις από το 2017 επίσης το Μητρό για την υποχρεωτική διαφάνεια για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μόνο τότε θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και να μας αντάξει των πολιτών ευχαριστούμε Μοντέλ Ε, πρέπει να ομολογήσω ότι η ανάγνωση της έκθεσης αυτής με θλίβει, διότι δεν περιέχει τίποτε το χειροπιαστό ή το συγκεκριμένο. Άδεια λόγια που ε, ε, επαναλαμβάνονται, χορεύουν γύρω-γύρω σε ένα τελείωτο βάλς χωρίς κανένα ρεφρέν. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε ότι γύρω από τη συμφωνία για τη διαθεσμική συμφωνία Έχουμε απόλυτη αδιαφάνεια. Βλέπουμε, α πούμε, την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Πώς προστατεύονται κοινωνικά οι Γάλλοι εργαζόμενοι και οι ίδιοι οι Γάλλοι πολίτες. Δεν βλέπω η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να θέλει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ε, πολιτών και των λαών, αλλά μόνο τα ε, άκρος φιλελεύθερα ε, συμφέροντα και τα συμφέροντα των πολυεθνικών. Δεν έχει νόημα η Ευρώπη αν δεν νομοθετούμε καλύτερα, αλλιώ να μην νομοθετούμε καθόλου. Θα πρέπει τα θεμελιώδη δικαιώματα του κάθε λαού, όπω θα έχει προβλέψει στην νομοθεσία του, να προστατεύονται με την ευφύ συνεργασία όλων των κρατών μεταξύ του. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει ε, μια ε, έγκυρη νομοθετική διαδικασία στα πλαίσια της δημοκρατίας. Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, Υπουργέ. Πρόκειται για μια πρώτη συμφωνία από το 2003 και ήρθαν αυτό το χρόνο. Εν γέννη, η νομοθεσία θα πρέπει να εκφράζει μια πολιτική βούληση για ρύθμιση κάποιων τομέων κατά τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο. Η νομοθεσία όμως δεν προκύπτει τυχαία. Πρέπει να διατυπώνεται με όσο δυνατόν περισσότερη περίσκεψη. Αυτή είναι μια διαδικασία χάραξης πολιτικής. Η νομοθεσία και αυτό είναι σαφές νομίζω ότι μέχρι τώρα συζήτηση, πρέπει να αποφεύγει τα, τα άκρα που είναι και η υπονομοθέτηση και η υπερνομοθέτηση. Άρα πρέπει να γίνεται ευρύτατη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και όχι μόνο με αυτούς που θα είχαν τις περισσότερες δυνατότητες για άσχεση πιέσεων μέσω των ομάδων των λόμπι. Πρέπει να αναγνωριστούν τα συμφέροντα των πάντων και των πιο δυνάμων πάνω από όλα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Φερρυπίν. Κάθε χάραξη πολιτικής προκύπτει από μια πολιτική επιλογή με νομικό αποτέλεσμα και έχει βέβαια και η υλοποίηση της νομοθεσίας, η εκτέλεση της, τη δική της σημασία. Πάντα πρέπει να δείχνουμε ευαισθησία στα θέματα αυτά και οι πολιτικοί πρέπει να χαράζουν πολιτική για να αντιμετωπίσετε κάθε πιθανό πρόβλημα. Σε έναν ιδεώδη κόσμο, καλύτερη νομοθεσία θα πρέπει να αποβαίνει σώφερος κάθε πολίτη της Ευρώπης και στην Ιευδία την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Ευχαριστώ, Μπρεσό. Grazie Presidente. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συνυπογραφή αυτή τη διοργανική συμφωνία είναι εξαιρετικό νέο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην φάση αυτή τη κρίση, όπου τα όρια αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα διάφορα θεσμικά όργανα μετακινούνται ή και εξαφανίζονται. Θέλω επίση να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μα, την Πρόεδρο Χούμπνερ, αλλά και τον σκιώδη εισηγητή Ρίτσερ Κόρπο και του τρει διαπραγματευτέ που εργάστηκαν για την επίτευξη μια θετική συμφωνία. Πιστεύω πω αυτή είναι καλή συμφωνία επιφέρει τροποποιήσεις που καθιστούν πιο ενήμερη την προηγούμενη συμφωνία του 2003. Ο διάλογος με του κοινωνικού εταίρους και τι μικρομεσαίες επιχειρήσει θα διατηρηθεί και θα αναπτυχθεί καθώς και η συμβολή τους θα ληφθεί περισσότερο υπόψη στη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, κυρίως και ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος των πράξεων θα αξιολογείται στη διάρκεια της ίδιας διαδικασίας. Επιπλέον, σε αυτή τη νέα συμφωνία εγγυάται την μεγαλύτερη διαφάνεια στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και το Ευρωκοινοβούλιο αποκτά μεγαλύτερο βάρος στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού, πράγμα που ζητάμε εδώ και καιρό. Θεωρώ λοιπόν πως είναι καλή η συμφωνία, αντιπροσωπεύει σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση, αν όχι της περισσότερο στενής ένωσης, αλλά της περισσότερο στενής ε, επαφής ανάμεσα στα ζωθεσμικά όργανα. Από αύριο θα πρέπει να ξεκινήσει η ισχύς λοιπόν εκείνη τη συνενέση. Καλύτερο είναι να νομοθετου... νομοθεσία σημαίνει καταρχάς να αποσύρουμε από το έδρανό μας και από το μυαλό μας τη σημαία της χώρας μας ο καθένας και να βάλουμε στη θέση της τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενος ομιλητής Βαζντόφσκι. Πρόεδρε, ευχαριστώ δεν είμαι οπαδός των ε, θέσεων που ακούστηκαν νωρίτερα, ωστόσο μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος σε ένα βαθμό για μια πιο λιτή νομοθεσία όπως φαίνεται να προκύπτει από την ε, συζήτηση. Θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση κάθε τμήματος της ε, διαδικασίας της νομοθετικής των συνεπειών και βέβαια σε σχέση με την ανταγωνιστικότητά μας. Υπάρχει βέβαια η αντίφαση, είτε επικουρικότητα, είτε κάτι το οποίο δεν μπορώ να δεχθώ 100% κόστος της αποτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό αποτελεί πρόσκληση προς κεντρική οργάνωση και υπερπαραγωγή νομοθεσίας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην πλάστικα στην επικουρικότητα να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο μέσα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι θα πρέπει και το ίδιο το Κοινοβούλιο να εισαγάγει στον κανονισμό του την αρχή τη επικουρικότητα, να μιλάει το ίδιο για επικουρικότητα. Ναι, λοιπόν, προ την ε, συμφωνία, αλλά όχι με τόσο ενθουσιασμό. τελικά Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Εγώ του Ναντίον ήμουν ενθουσιώδη υποστηρικτή. Επρόκειτο για μία από τι προτεραιότητε με τι οποίε μπήκα ω Ευρωβουλευτή στο Κοινοβούλιο και είχαμε τη συζήτηση αυτή με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαντς και το 2014 με τις προτεραιότητες. Καταλαβαίνω ότι είχατε πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες και, και φιλοδοξίες όπως και εγώ και πολλοί άλλοι πιστεύω. Αλλά από την άλλη υπήρχαν και άλλοι που είχαν χαμηλότερες φιλοδοξίες και έτσι τελικά βρισκόμαστε ενώπιον ενός συμβασμού που εσείς θα πείτε ότι είναι μισογεμάτο το ποτήρι, ίσως περισσότερο από μισό θα έλεγα. Μια συμφωνία πάντως καλή και νομίζω μπορούμε να το γεμίσουμε το ποτήρι χάρη στην υλοποίηση της συμφωνίας με τον διαπραγματευτή μας Γκίφερ Χόφστατ και μακάρι να ήταν εδώ παρόν να ακούσει αυτά που έχω να του πω αλλά πιστεύω ότι έκανε πολύ καλή δουλειά και θα τα πω έστω και απουσία του. Έχουμε νομίζω μια συμφωνία που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε σήμερα έτσι ώστε όπως είναι παρόντερα να γεμίσουμε το ποτήρι. Ένα παράδειγμα θα δώσω. Να, ένα παράδειγμα επί παραδείγματι, να σβήσω και λίγο από το φόρτο αυτή της ε, πλεοναστική φράση. Το γραφειοκρατικό, το διοικητικό βάρος. Ακριβώς εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να δείξει ικανότητα και θάρρος η Επιτροπή ώστε να υποδεικνύει ποιος προτείνει τι σε κάθε τομέα και πώς θα συμπεριφέρονται τα κράτη-μέλη. Αυτό ακριβώς νομίζω μπορεί να δείξει χάρη στις προτάσεις, τις προτάσεις που θα προχωρήσουν, τα νομοθετήματα ώστε να μην υπάρχει αυτή η ε, υπερβολική νομοθέτηση. Και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει το εργαλείο να φέρουμε απτά αποτελέσματα. Σε ευχαριστώ θερμά και νομίζω ότι εδώ θα κρυθούμε από το πώς θα υλοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Χίμπνερ, στην έκθεσή σας έχετε επισημάνει την ανάγκη να υπάρχουν περισσότερο συγκεκριμένες διατάξεις για τη διαφάνεια όλων των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τις κατεξοδότητες πράξεις Μάλιστα, στο ίδιο, αποτέλε... στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε πριν από δύο εβδομάδε και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Είναι απαραίτητη για την καλή εφαρμογή τη νομοθεσία η καλή συμμόρφωση. Η διοργανική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία επιτρέπει μια πιο διαφανή λοιπόν και πιο ε, εύρυθμη συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τώρα στα μισά του δρόμου. Να εξηγήσω ότι ενώ η εξακολούθηση για την καλύτερη νομοθεσία είναι να υπάρξει καλύτερη διοικητική μηχανή. Είχα την τύχη να ετοιμάσω ένα σχέδιο κανονισμού για ανοιχτό, διαφανή και ελεύθερο διοικητικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παρουσιαστεί και εδώ του ερχόμενου μήνε. Ο Υπουργό γνωρίζει πολύ καλά αυτό το εγχείρημα, διότι είναι πρώην μέλο ε, ε, του σώματο. Ξέρετε λοιπόν ότι οι καλύτερε και απλοποιημένε διοικητικέ διαδικασίε μπορούν να ε, βελτιώσουν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ αφήσουμε προσπαθειών για να πετύχει καλύτερη νομοθεσία και απλοποίηση τη διοικητική μηχανή του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κυρίω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει την αλία, τη γεωργία, το εμπόριο, έχετε την νομική Πριτανία και έχετε τους ε, πρωθυπουργούς, τους πρωθυπουργούς ε, στην πρώτη γραμμή. Θέλετε ανοιχτά και ολοκληρωμένα σύνορα, θέλετε έναν στρατό. Και ακόμη και όταν αποτυγχάνει το νόμισμά σας δεν το βάζετε κάτω. Θέλετε περισσότερη διαφάνεια ενώ η οικονομία σας κλειδονίζεται. Λίγοι δωρεάν, ε, κάποιες δωρεάν συμβουλές. Αν θέλετε καλύτερη νομοθεσία, σταματήστε να νομοθετείτε. Όλα αυτά που ανέφερα είναι αρμοδιότητες των κυρίαρχων εθνικών κρατών. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το ε, τόπο. Πολύ σύντομα το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ελεύθερο και θα πάρει πάλι τι αρμοδιότητε πίσω στα χέρια του από αυτήν την Ένωση. Τόσο το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριο Πίπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. πιστεύαμε κάποιους από τους προοραλήσαντες, σήμερα έχουμε έρθει σε μια μεγάλη ρήξη. Ε, όχι λοιπόν, αν κοιτάξουμε την πρόταση της Επιτροπής, μέσα από τον τριμερή διάλογο πολλά χάθηκαν. Βλέπει ο, πρόεδρο, ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς μισογεμάτο το ποτήρι, ο, πρόεδρος Φερχόφστατ δεν είναι σήμερα εδώ. Θετικά πάντως μπορούμε να το κρίνουμε. Ακολουθεί και το Συμβούλιο την ιδέα της κατάρρησης της γραφειοκρατίας. Περισσότερη ανεξαρτησία προς την αξιολόγηση της ποιότητας και των συνεπειών. Θετικά νομίζω μπορούμε να κρίνουμε και την ανάγνωση του Κοινοβουλίου με την έκθεση Χιούμπνερ και θέλω να ευχαριστώ ρητά τους κυρίους Βερχόφστατ και Χιούμπνερ. Αλλά πάντως η Επιτροπή ήθελε μια πιο σαφή υποχρέωση λογοδοσίας για την υπερβολική νομοθέτηση. Γιατί λοιπόν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποδυναμώνουν τις σχετικές διατάξεις. Γιατί δεν θέλουν τις ευθύνες. Για το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο απεισχνάζουν αυτή την πρόταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έναν ετήσιο κατάλογο με τις νομοθετικές προτάσεις τα δηλαδή Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο απεισχνάζουν και ε, είναι ο αποδεπομπαίο τράγος τη Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται λοιπόν να μιλήσουμε περισσότερο για διαφάνεια, αλλά τα λόγια αυτά, οι φράσει αυτέ χάθηκαν. Κρίμα. Κρίμα διότι θα μπορούσε περισσότερο να καταλάβει ο πολίτης ποιος είναι υπεύθυνο σε ποια φάση για την εισαγωγή τίνος νομοθετήματος στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Και έτσι θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μπορεί να ήταν πιο γεμάτο το ποτήρι, κυρία Πρόεδρε, αλλά θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Ευχαριστώ. Κυρία Κάουφμαν, η ίδια οργανική συμφωνία για την οποία σήμερα, ε, αύριο θα ψηφίσουμε. Είναι μια καλή συμφωνία, αποτελεί μια καλή βάση για τη συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ταυτόχρονα αποτελεί και καλό νέο για τον πολίτη της Ευρώπης. Γιατί, Γιατί με τη συμφωνία αυτή καθιστούμε σαφές ότι δεχόμαστε με σοβαρότητα τις κριτικές, θέλουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο δράσης και λειτουργίας μας, θέλουμε να βελτιώσουμε την νομοθεσία και στοχευμένα να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία. Πριν να προχωρήσω θέλω να προσθέσω μια ακόμη πτυχή. Με την καλύτερη νομοθέτηση μπορούμε να έχουμε όχι απλώς μείωση του αριθμού του καθαρού αριθμού των νομοθετημάτων, γιατί δεν είναι θέματα περισσότερα ή τα λιγότερα νομοθετήματα, αλλά η ποιότητά τους. Όταν έχουμε να κάνουμε με ποιότητα περιβάλλοντος, προστασία του καταναλωτή, του εργαζομένου, τα ποιότητα, έλεγχο ποιότητα των προϊόντων. Αυτά τα περιμένει ο πολίτη και εδώ η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μπορούσαν να κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ, Βαν Μποσουίτ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Αύριο θα εγκρίνουμε κάτι που μοιάζει αυτονόητο. Προφανώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θέλουν καλύτερη νομοθεσία και απλούστερη. Χρειαζόμαστε νομοθεσία η οποία να μπορεί να υλοποιείται εύκολα και να μειωθεί το διοικητικό άχθος. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι φιλοδοξίες μας στέκονται στο ύψος των ε, περιστάσεων. Οι προσπάθειες ε, του κυρίου Φερχόφστατ που είναι υπέρ της Ευρώπης δεν ε, αντικατοπτρίζονται δυστυχώ και στην πραγματικότητα όπω θα έπρεπε με του εκπροσώπου που έχουμε εδώ. Ε, δυστυχώ ο κ. Φερχόφστατ αγωνίζεται μόνο του. Εδώ λοιπόν η έλλειψη διαφάνεια ε, στην όλη διαδικασία δεν έχει εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ε, είναι η παρακαταθήκη μα για το μέλλον. Δηλαδή να πούμε αντίο στην παλιά Ευρώπη και να χτίσουμε επιτέλου την καινούρια. Ευχαριστούμε. Άντερσον. Πρόεδρε, αυτή η διοργανική συμφωνία μεταξύ Επιτροπή Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, εκπονεί νομοθεσία στο μέλλον έχει κάποια θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία. Το πιο σημαντικό όμω είναι ότι οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει πλέον να παραλύουν την νομοθετική διαδικασία. Δηλαδή, ε, το ερώτημα είναι θα υπάρχουν μήπως υπερβολικά πολλές μελέτες αντικτύπου. Γιατί είπαμε να αποφύγουμε το υπέρμετρο στοιχείο στην νομοθεσία. Βεβαίω είναι καλό να αναλύουμε, να αναλύουμε τον αντίκτυπο των προτέρων. Είναι κάτι θετικό. Όμω πρέπει να σκεφτούμε και το κόστο για του επιμέρου παραγωγού, λόγω χάρη. Οι εταιρείε που παράγουν επικίνδυνα χημικά προϊόντα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το κέρδο από το να μην έχουμε χημικέ ουσίε ε, στην αγορά είναι σημαντικό. Πάνω απ' όλα. Οπότε, εάν έχουμε υπερβολικά πολλέ μελέτε αντεκτύπου, μπορεί να παραλύσουμε την όλη διαδικασία και όχι να πετύχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε, Σιέφκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Ε. συνάδελφοι, θα ήθελα να συμφωνήσω με όσο από σας είπατε ότι δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα των συμφωνιών, των διποματεύσεων και την διοργανική συμφωνία. Ωστόσο, Μόνο αυτό καταφέραμε να είναι το αποτέλεσμά μας, ε, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Θα μπορούσαμε όμως ε, αυτή τη συμφωνία να την καταψηφίσουμε. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, θα περάσει, διότι είναι θεμελιώδου σημασία η συνεργασία μας να συνεχιστεί. Να σχολιάσω ότι οι διαπραγματεύσεις παρόλα αυτά δεν πήγαν όπως θέλαμε και ότι πέραν των όσων περιέχει η διαθεσμική αυτή συμφωνία, προσδοκούμε επιτέλους αυτή η συμφωνία να γίνει πλήρως σεβαστή και από τα τρία θεσμικά όργανα. Στο Κοινοβούλιο κάθε χρόνο συζητάμε την, ιδίως την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, τα του κοινοτικού δικαίου, τη δημιουργία νέων μηχανισμών, για να μπορούμε να σεβόμαστε περισσότερο το κοινοτικό δίκαιο. Όμω, για την ε, αγαστή συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, μην ξεχνάμε ότι δεν αρκεί μόνο αυτό για να έχουμε καλύτερη νομοθεσία. Πρέπει να παρουσιάζονται καλύτερε προτάσει με ε, πιο εύστοχα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Άρα δεν αρκεί να έχουμε μόνο καλούς στόχους και είναι κρίμα παρά τις πολλαπλές μας απόπειρες, προσπάθειες και την αιμονή της δικής μου ομάδας προς αυτό το στόχο τελικά με τις μελέτες αντικτύπου να μην έχουμε αυτά που είχαμε επιδιώξει ακόμη και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόσχεται ευρύτατες διαβουλεύσεις. Και ε, εντός μισού λεπτό θα ολοκληρώσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλά για τη μελέτη αντικτύπου για τους κτηνοτρόφους και για την κατάσταση της κτηνοτροφίας. Ε, Ποιε είναι οι διαβουλεύσει που ε, διοργανώθηκαν ή κρεπατόμαστε μεταξύ μα ή δεν εργαζόμαστε για κοινό σκοπό. Ευχαριστούμε, σύχτα. Ευχαριστώ. Η αύξηση τη αποτελεσματικότητα είναι σημαντική για την βελτίωση τη οικονομία, για την δημιουργία ευημερία και θέσεων απασχόλησης. Θέλουμε λοιπόν να αρθούν τα γραφειοκρατικά άχθη και να μειωθεί το κόστο που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσει και οι διοικητικέ υπηρεσίε όταν προσπαθούν να συμμορφωθούν με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτή η νέα συμφωνία θα πρέπει να δεσμεύει και το Κοινοβούλιο και τα 28 κάτι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που από κοινού θα πρέπει να συνεργαστούν για την καλύτερη νομοθεσία. Μόνο έτσι θα πετύχουν του στόχου μα. Όμω δεν μπορούμε να πάμε μακρύτερα. Ε, τον περασμένο μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Αρχική Κατόνια Κυβερνήσεων αποσχέθηκαν ένα τομέα εξέταση για να αρθεί το περιττό κόστο που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτέ και επιχειρήσει. Οι οικονομίε μα δεν μπορούν πλέον να πληρώνουν για άδειε υποσχέσει. Επίτροπε, κράτη-μέλη, κοινοβούλιο, ας εργαστούμε σκληρά, ας ανασκουμποθούμε για να πετύχουμε αποτελέσματα. Σφαβόντα. Ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Εγώ μιλώ εδώ ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, Νομικών Υποθέσεων, τις οποίες ε, καθήκον μεταξύ άλλων είναι να βελτιώσει την νομοθετική διαδικασία. Είναι σίγουρα θετικό ότι έχουμε μια νέα διοργανική συμφωνία. Ωστόσο, το Ευρωκοινοβούλιο ε, ήδη στο παρελθόν έχει ορίσει κάποιες ε, παράγοντες που εν μέρη έχουν ήδη εφαρμοστεί. Ας πούμε, η αξιολόγηση αντικτύπου είναι πολύ σημαντική υπόθεση για την εκτίμηση της ποιότητας της νομοθεσίας. Τέτοιες αξιολογήσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε νέα νομοθεσία δεν προκαλεί υπερβολικό δι, ε, διοικητικό άχθος για τους χρήστες. Ε, Μία από τις πρώτες μας προτεραιότητες λοιπόν είναι αυτή η αξιολόγηση αντικτύπου και δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Επίσης προβλέπονται νέα βήματα όσον αφορά τις εφαρμοστικές και τις κατεξοδότηση πράξεις. Μόνο μετά από κάτι τέτοιο θα είναι πιο ολοκληρωμένη η συμφωνία. Τέλος, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα παρακολουθήσουμε την εφαρμογή του συνόλου αυτής της συμφωνίας, γιατί μόνο έτσι θα είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε ένα λειτουργικό μέσο που θα παίξει το ρόλο του. Γι' αυτό και η Επιτροπή Νομικών μαζί με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα παρακολουθούμε στενά ε, την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας μέσω εκθέσεων ίδιας πρωτοβουλίας και μέσω κοινή μας συνεργασίας. Ευχαριστώ. Επόμενος ο κύριος Ράντεφ. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω πως θα μπορούσαμε να είχαμε καταλήξει σε καλύτερη συμφωνία. Το κείμενο που έχουμε είναι αποδεκτό, αλλά δεν είναι επαρκές. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε πιο απλές νομοθεσίες παρά να αυξάνουμε τη γραφειοκρατία για τους Ευρωπαίους πολίτες ή για τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Ε, το μέτρο, η μέτρηση του γραφειοκρατικού άχθους θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε τις εργασίες της Ένωσης και να τονίσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει, γίνει να... θα πρέπει επίσης να γίνει ε, μια διάκριση ανάμεσα στο φόρτο που προκύπτει από τα νομοθετήματα των Βρυξελών και τα νομοθετήματα των κρατών, των εθνικών ε, νομοθετών, έτσι ώστε να μην κατηγορούνται πάντα οι Βρυξέλλες. Επίσης, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στις επιπτώσεις των νέων νομοθεσιών στην ανταγωνιστικότητα. Η ετήσια μελέτη για τον διοικητικό φόρτο και οι αξιολογήσεις αντικτύπου θα μας επιτρέψουν να μετρήσουμε τον αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ελπίζω πόσο οι διατάξεις αυτής της συμφωνίας θα εφαρμοστούν σωστά και θα συμβάλλουν σε καλύτερη ευρωπαϊκή νομοθεσία, νομοθεσία ενημερωμένη και ποιοτική. Ευχαριστώ. Τόμασιτς. Σας ευχαριστώ. Σημερίζομαι τις συστάσεις της εισηγήτριας αλλά και την ανησυχία της όσον αφορά τον αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η βάση της ευρωπαϊκής οικονομίας και δίνουν δουλειά στο 80% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Κάθε υπεύθυνος νομοθέτης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μικρομεσαίων. Από αυτό εδώ το σώμα ζητάμε την ε, Αξιολόγηση επίση του αντικτύπου τη κάθε νομοθεσία για την ισότητα των φύλων. Οι ίδιε οι μικρομεσαίε επιχειρήσει εξασφαλίζουν πάλι ένα μήνυμο με ισότητα. Είναι εξαιρετικά σημαντικέ. Όταν ε, πρόκειται λοιπόν για νομοθεσίε και νομοθετικέ πράξει, η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ποσότητα και ελπίζω έτσι ότι θα μπορέσουμε να, φτιάξουμε, να φτάσουμε σε μια πραγματική γιγιοτίνα ρυθμιστική όπου θα ακυρώνονται οι περιττέ νομοθεσίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο έτσι οι επιχειρήσει μα να μπορέσουν να ωφεληθούν από την ενιαία αγορά και να προσφέρουν δουλειά σε περισσότερους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στο Κατζέι. Θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο σε όλους, αλλά θα πρέπει να τηρήσετε το ένα λεπτό. Πρώτος είναι ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θετικό σήμα απέναντι σε αυτή τη διοργανική συμφωνία και θεωρώ πως είναι μια καλή βάση για να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν οι σχέσεις και η διαφάνεια ανάμεσα στα θεσμικά όργανα με στόχο το καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πολίτη. Είναι καλό το να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων ε, διαθεσμική ε, για τις νομικές βάσεις και είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που υπάρχουν στη διαθεσή μας ώστε να νομοθετούμε σωστότερα αξιολόγηση αντικτύπου, δημόσια διαβούλευση, αναλύσεις έτσι ώστε η διαδικασία λήψη αποφάσεων να είναι ενημερωμένη και εμπεριστατωμένη. Θα πρέπει επίση να ανταλλάσσουν απόψει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ω νομοθέτε και αυτό είναι ένα βήμα μπροστά. Ωστόσο, θεωρώ πω πρέπει να γίνει βάθυνση ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, αμοιβαία πρόσβαση στις πληροφορίες της Ένωσης, ώστε να είμαστε σίγουροι για την ισότητα πρόσβασης στη διάρκεια της διαβούλευσης. Ε, και έτσι θα εγγυηθούμε και την αρχή της σωστής και πιστής συνεργασίας. Ευχαριστώ. E Ευχαριστώ. Η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχει να κάνει με, ε, μοιάζει με το ποδήλατο. Αν κανεί σταματήσει να πατάει τα πόδια του στο πετάλι και να κινεί το ποδήλατο, φαίνεται σαν να πρόκειται να καταρρεύσει. Εδώ λοιπόν, με τόσε εκατοντάδε νομοθετικέ πράξει, φαίνεται ότι κανεί δεν μπορεί να μα δώσει τον συνολικό ακριβή αριθμό. Το ίδιο και οι ποδηλάτε ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι 3.000 υπάλληλοι, και με όλα αυτά, ε, καλό θα είναι να θυμόμαστε τι είχαμε συμφωνήσει τη στιγμή ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να νομοθετούμε όταν είναι χρήσιμο και όταν στο, ε, και μόνο στο βαθμό που είναι χρήσιμο. Αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε πότε πότε στην ε, ζωή που διάγουμε εδώ, ό,τι και γνώμη και αν έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Πρέντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε ε, για τις προτάσεις αυτές. Καλύτερη ε, νομοθεσία, διοργανική συμφωνία είναι τα βασικά στοιχεία που θέλω να σχολιάσω. Καλύτερη νομοθεσία λοιπόν. Για ποια... Με ποια κριτήρια και για ποια συμφέροντα. Από ό,τι βλέπουμε η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μάλιστα τα συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων θα καθορίζουν τις ευκαιρίες ε, της πρόοδου της συνομοθεσίας. Εδώ τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα ίσως να μην μπορούν καν να φτάσουν να βελτιώσουν τη διαβίωση των λαών της Ευρώπης. Επίσης υπάρχουν σοβαρές ε, δυσκολίες για την δημοκρατικότητα των διοικητικών διαδικασιών. Χρειάζεται, φαίνεται να υπάρχει περισσότερη συγκέντρωση των εξουσιών στην Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και επίσης η δυνατότητα παρέμβασης των συνομοθετών, ιδίως των βουλευτών, να περιορίζεται. Τρίτον, η διαφάνεια φαίνεται ότι παρά τις καλές μας προθέσεις ως προς αυτό το θέμα δεν υπάρχει αντιστοιχεία με την πραγματική ζωή. Τα έγγραφα συνεδριάσεων και δημοτεύσεων δεν αποκαλύπτονται για πολλούς ε, λόγους εμποδίζοντας την διαφάνεια των ε, διάφορων διαδικασιών. Στη, στο σκοτάδι υπογράφονται και ακριβώς αυτό δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ευχαριστούμε ο κ. Καστάλντο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ερώτηση που θέσαμε στους εαυτούς μας στην αρχή αυτής της συζήτησης είναι αν θέλουμε το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Αυτό μου φαίνεται, αλλά α, αναλόγως με την οπτική γωνία του καθενός και τα δύο μπορούν να ισχύουν. Εγώ θα λέγω ότι είναι περισσότερο μισοάδιο. Βεβαίως έγιναν κάποια βήματα πρόοδου, λόγω χάρη ακριβώς το θέμα του χρονοδιαγράμματος ή οι μελέτες αντικτύπου. Όμως μετά θα πρέπει να δούμε ποιος θα τα αναλάβει όλα αυτά. Ποιο θα τα κάνει αυτά για λογαριασμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, βεβαίω και αυτό είναι ε, προσφυλέ στο κίνημα το οποίο εκπροσωπώ. Όμω δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουμε προ όφελο μια νομοθεσία που θα ελαφρά, ελαφρύνει το διοικητικό του άχθο, να δημιουργήσουμε ένα δόριο ύπο που ουσιαστικά θα ε, πλήξει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών που και αυτοί εκπροσωπούν ε, εξυπηρετώντα τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών. Επίση και για διαδικαστικά και έχουμε επικρατικά σχόλια. Δηλαδή, δεν φαίνεται τα θέματα που το, Ευρωβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να θέσει, να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, αλλά και για τη διαφάνεια των τριμερών διαλόγων. Δεν αρκεί να ξέρουμε εκ των υστέρων τι υπόθηκε, αλλά για να ακολουθήσουμε τι προδιαγραφέ των συνθηκών θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία να είμαστε διαφανεί. Δεν είναι κάτι που το δημοτεύομαστε αυτό. Ο κύριος Συναντινός. Κύριε Πρόεδρε, η νέα διοργανική συμφωνία για την βελτίωση τη νομοθεσία είναι ένα γράμμα κενό νόμου. πρωτοετή φοιτητή τη νομική θα μιλούσε για κενό δικαίου. πολάκη η γραμματική ιστορική τελεολογική και συστηματική ερμηνεία του δικαίου τη ένωση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τι αρχέ τη αναλογικότητα και επικουρικότητα καθώ και την ασφάλεια δικαίου. τα παραδείγματα πολλά και τα γνωρίζουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα όταν για παράδειγμα η επιτροπή αποστέλει νομοθετικέ πράξει ή οδηγίε μη λαμβάνοντα υπόψη τις παρατηρήσεις των διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών ακόμα και μετά το πέρας δύο αναγνώσεων. πολλές και οι περιπτώσεις μη μεταφοράς του κοινοτικού δικαίου στα αντίστοιχα εθνικά. η νομική επιστήμη δεν είναι θετική επιστήμη διότι τα πορίσματά της δεν μπορούν να επαληθευθούν με πειράματα. οι θεσμοί δυστυχώς έχουν καταντήσει τους πολίτες της ένωσης πειραματόζωα εσφαλμένων οικονομικών κυρίως πολιτικών και νομοθετημάτων. ευχαριστώ. Χορεγκούι, παρακαλώ. Εγώ θέλω να συμφωνήσω με αυτή τη ε, διαργανική συμφωνία και να θυμίσω δύο σημαντικέ πτυχέ, κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, να θυμίσω ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται μια διαδικασία στο Οικομισιόν να πρέπει να απαντήσει στι προτάσει που προέρχονται ε, από το Κοινοβούλιο. Η συμφωνία ορίζει τρει μήνε διορία μέχρι ότου η Οικομισιόν να δώσει απάντηση ή κάποια συνέχεια στι ε, προτάσει πρωτοβουλία που προκύπτουν προκύπτουν από, αυτή, από αυτό το σώμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί γνωρίζουμε ότι κάποιες, πολλές φορές οι εκθέσεις πρωτοβουλία που προκύπτουν από το Κοινοβούλιο πολλές φορές κοιμούνται στα σερτάρια των Κομισιών. Αυτή λοιπόν η διορία για απάντηση είναι πολύ σημαντική και κατά δεύτερο λόγο είναι σημαντική η υπόσχεση για περισσότερη δυνατότητα πρόσβαση στην ενημέρωση, στα έγγραφα και στην συμμετοχή των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, γιατί το να βελτιωθεί η σχέση ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα ευνοήσει και την νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριάς. Έχω κάνει συχνά κριτική στην Κομισιόν για τη γραφειοκρατία που έχει, για τη σύγκρουση συμφερόντων που παρουσιάζει ως μέλος της Τρόικας και ως θεματοφύλακας των συνθήκων. Αλλά θέλω να πω κάτι και να απευθυνθώ στο σώμα. Έχει δει το Προεδρείο τι νέα γραφειοκρατία έχει φάλει με τον νέο τρόπο πρόσληψης των τοπικών συνεργατών των βουλευτών. έχετε ασχοληθεί πραγματικά με το τι γραφειοκρατικό τέρας έχετε δημιουργήσει. εάν κάποιος θέλει να προσλάβει κάποιον με τηλεεργασία ο οποίος δεν μένει στην αθήνα φερρυπίν και μένει στη θεσσαλονίκη δεν μπορείς να τον προσλάβεις με σύμβαση αορίστου χρόνου διότι πρέπει να έρθει να εγκατασταθεί στην αθήνα και σου λέει να τον προσλάβεις με σύμβαση ελευθέρων, ε, παροχής ελευθέρων υπηρεσιών. Πολύ απλά το ίδιο το Κοινοβούλιο με τη γραφειοκρατία που έχετε βάλει έχετε κάνει έτσι την κατάσταση που να μην μπορούμε ούτε να προσλάβουμε τοπικούς βοηθούς ούτε να αναθέσουμε υποθέσεις. Τεράστια γραφειοκρατία. Ένα έγγραφο που είχε πέντε ε, σελίδες το κάνατε πενήντα σελίδες. Λοιπόν, πριν κάνουμε κριτική στην Κομισιόν, ας αποφασίσει και το Κοινοβούλιο να μαζέψει τη γραφειοκρατία που έχει κάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι γνωρίζουν ήδη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δημοκρατικός θεσμός. Δεν μπορεί να είναι δημοκρατικός ένας θεσμός που απαιτεί την πληρωμή του χρέους σε αντίθεση με τη διατήρηση των δημοσίων υπηρεσιών που υποχρεώνει τους εργαζόμενους να εγκαταλείψουν τα εργαστικά τους δικαιώματα που αρνείται να ανοίξει τα σύνορά της στους πρόσφυγες που φεύγουν από πολέμους που ήδη τροφοδοτεί. Ε, Ποιο ξέρει, ίσω με διαφορετικέ πλειοψηφίε να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αν ήταν οργανωμένοι, δηλαδή οι εργαζόμενοι και μπορούσαν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά του απέναντι στι ολιγαρχίε. Όμω με τέτοιε προτάσει όπω η σημερινή αρνούμεθα τέτοια δυνατότητα, γιατί αποσύρεται από το Κοινοβούλιο η δυνατότητα να αποφασίζει ω αντιπροσωπευτικό ε, όργανο της Λαϊκής Βούλησης. Αφήνουμε να αποφασίζει η μη εκλεγμένη γραφειοκρατία της Κομισιόν. Πρόκειται για μια ε, ε, μια για μας μάλλον η νομοθεσία ε, δεν είναι ένα συμπλήρωμα των συμφερόντων της αγορά. Δεν μπορούμε να τα καταλήψουμε ως κοινοβούλιο την νομοθετική διαδικασία. Ο κύριος Τίμερμαν τώρα. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε μερικά σχόλια για τα όσα άκουσα. Πρώτα απ' όλα, δεν δύναμε να αντιληφθώ πώς μπορεί κανείς να ισχυρίζεται ότι το να κάνουμε, να λαμβάνουμε μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστά νεοφιλελεύθερη πολιτική. Εάν μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ώστε οι επιχειρηματίες αυτοί να μπορούν να ασχολούνται με τις επιχειρήσεις τους και να μην χρειάζεται να περνούν ώρες ατελείωτες σε επικοινωνία με τη διοίκηση, θα μπορούσαν να προσλάβουν και επιπλέον προσωπικό. Πώ μπορεί να είναι αυτό λογικό, εάν μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερε θέσει εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα από τι μικρομεσαίε θα ξεκινήσουμε. Είναι το καλύτερό μα ατού. Το πρόγραμμα αυτό, αυτή η συμφωνία, μα επιτρέπει ιδιαίτερα να εστιαστούμε στι μικρομεσαίε. Γιατί γιατί δεν μπορούν μόνες τους να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους όπως οι μεγάλες μπορούν μέσα σε αυτό το, σε αυτό το θόλο των Βρυξελών. Γι' αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους μικρομεσαίες. Δεύτερον, κύριε Τζιχόν, ε, εξανέστησαν οι πράσινοι. Εξανέστηκε ο κύριος Ντουρό ο ίδιος, γιατί θεωρεί ότι μειώνουμε τις κοινωνικές προδιαγραφέ, τις περιβαλλοντικές εγώ εκάλεσα, εγκάλεσα την ομάδα του τρεις φορές να μου δώσει, πολλές φορές να μου δώσει τρία παραδείγματα συγκεκριμένα όπου προτάσει Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάθμισαν τις κοινωνικές περιβαλλοντικές προτεραιότητε. Και δύο και ένα θα μου έφτανε. Αλλά όχι. Ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν πριν εκνευριστεί καλύτερα να συνομιλεί και με τους συναδέλφους ομάδας του για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Και εν τέλει επιτρέψτε μου δεν παραλάβω σαφέστατα ότι για μένα αυτό είναι η απαρχή μιας διαδικασίας. Ο τρόπος με τον οποίο θα την υλοποιήσουμε τη συμφωνία αυτή θα δείξει το τι μπορούμε να πράξουμε, εάν δηλαδή είμαστε ικανοί να έχουμε καλύτερη νομοθεσία ή όχι. Δεν πρόκειται μόνο για λιγότερη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται και για μια ορθολογική ρύθμιση κατά τρόπο οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά ανεκτό και βιώσιμο, μείωση της γραφειοκρατίας και εξέβρεση κοινή λύση. Αυτό σημαίνει επίση καλύτερη νομοθεσία. Και είμαι υπερήφανο για το γεγονό ότι με αυτή τη συμφωνία. Επαναλαμβάνω για μια φορά ότι θα ήθελα να είχαμε επιτύχει περισσότερα ακόμα. Αλλά πάλι αυτό είναι η συνένεση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, των διαφορετικών πολιτικών θεωρήσεων στην υπόθεση αυτή και συνιστά νομίζω τη βάση για μια πραγματικά καλύτερη νομοθεσία. Με έλεγχο απόλυτο από τον έξω κόσμο θα είμαστε πολύ πιο διαφανείς, πολύ πιο ανοιχτοί και θα περιλαμβάνουμε και τους άλλους. Ιδιαίτερα με τις πλατφόρμες που θα δημιουργήσουμε θα επιτρέψουμε την παρακολούθηση και την νέα ορμή στην υπόθεση αυτή ώστε να μην επιβαρύνονται κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από περί την νομοθεσία και γραφειοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα θα λάβει η Υπουργό Σένις Πλάσετ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που σας μίλησατε για τη σημασία της αξιολόγησης των συνεπειών. Βεβαίως είμαι και εγώ πεπισμένη ότι θα ενισχυθεί αυτή η διαδικασία αξιολόγησης των συνεπειών και είμαι πεπισμένη ότι θα επιτρέψει ε, στα θεσμικά όργανα να αξιολογούν καλύτερα την υλοποίηση σε πρώιμο στάδιο των συνεπειών της ε, νομοθεσίας βέβαια αυτή η αξιολόγηση συνεπειών δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζει το ρόλο των συνομοθετών είτε αυτό το κοινοβούλιο είτε το συμβούλιο θα πρέπει μόνο να ε, συμβάλλει σε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και έτσι θα συμφωνήσω με τους ομιλητές που τοποθετήθηκαν υπέρ των, των αξιολογήσεων συνεπειών εμείς ως συνομοθέτες εν τέλει θα πρέπει να λαμβάνουμε τις πολιτικές αποφάσεις Όσο καλύτερη όμω είναι η αξιολόγηση των συνεπειών, τόσο καλύτερε και οι πολιτικέ αποφάσει που θα ακολουθήσουν. Ο κύριο Πίπερ αναφέρθηκε στο ζήτημα τη ε, περί τη νομοθεσία. Είναι σαφέ νομίζω στο κείμενό μου και καταγράφεται ιδιαίτερα ο ρόλο των θεσμικών οργάνων ως προς την αξιολόγηση και την υλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σημασία έχει να έχουμε μια απόλυτα σαφή εικόνα όλοι μας για τις πτυχές της εθνικής νομοθεσία που μπορεί να έχουν ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκό χαρακτήρα και ποιε θα πρέπει να παραμένουν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό νομίζω είναι σαφώ διατυπωμένο στη συμφωνία. Νομίζω ότι ακούστηκαν ε, οι επιθυμίες και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και οι θέσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων που έχουν και ιδιαίτερο ρόλο στη διαδικασία της υλοποίησης. Ο κύριος Πίπερ ξέρω ότι θα θέλει να προχωρήσουμε περισσότερο προς την ε, αντιμετώπιση περί της νομοθεσίας αλλά ελπίζω ότι θα δεχθεί όπως είπε και ο Τίμερμανς, ότι το μισογεμάτο ποτήρι μπορεί και αυτό να είναι εύγευστο. Για την κυρία Τινόλφ και άλλους ε, η σημασία της ενίσχυσης της διαφάνειας και σε αυτό τοποθετήθηκα νωρίτερα, θα το τονίσω για άλλη μια φορά. Η Προεδρία των Κάτω Χωρών ξεκινάει με δύο σημαντικές διατάξεις στη συμφωνία το μητρό των κατεξουσιώτων συμπράξεων και την καταγραφή των νομοθετικών ε, πράξεων και πιστεύω ότι και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα προχωρήσουν προς την διακατεύθυνση για να ενισχυθεί η διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, νομίζω ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ξεκάθαρα μίλησε για το θέμα αυτό και συμφωνώ με την κυρία Βίκη ότι πρέπει να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας. Είμαι πεπισμένη ότι αυτό θα πράξουμε και πριν κλείσω, Πρόεδρε, θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω τους Γκίφερ Χόφστατ, τον Φραντ Τίμερμανς και τον Νίκολα Σμιτ από την Πρόεδρε του Λουξεμβούργου και την εισηγήτρια κυρία Χιούμπνερ τους συνεργάτες της, τους, τους είπα, στην Επιτροπή. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί και πρέπει να ε, δει τη συνεργασία των θεσμικών οργάνων. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Χιούμπνερ το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τα δύο θεσμικά όργανα, τα άλλα δύο θεσμικά όργανα που ήταν σήμερα μαζί μα. Να πω στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου, την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου που εκπροσωπεί την Ολλανδική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπεί ο Πρόεδρο Τίμερμαν, ότι του ευχαριστώ για την αφοσίωσή του στην υλοποίηση τη Διαθεσμική Συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία. Και Είμαι βέβαια ότι αν σε στενή συνεργασία προσπαθήσουμε αυτή την πραγματική υλοποίηση και έχουμε μια υφή υλοποίηση, δεν θα χρειαστεί να κάνουμε αυτήν την παραπάνω εξαντλητική προσπάθεια, όπως είπατε κι εσείς, Αντιπρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για την καλύτερη νομοθεσία και όπως και εσείς προσπαθήσατε να το περιγράψετε, πρέπει να πάμε πέραν των όσων λέει το χαρτί και να δεσμευτούμε γι' αυτό. Το Συμβούλιο έχει αρχίσει τη συζήτηση για την υλοποίηση και θα βεβαιωθεί για την συνέχιση, την εξακολούθηση των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό για μα είναι πολύ ευχάριστα νέα. Αλλά για μα εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο σημαντικό είναι να προχωρήσουμε για την καλύτερη νομοθεσία, ενώ θα σεβόμεθα την ποιοτική αγαστή συνεργασία μεταξύ των ε, συνομοθετών. Έχουν αναλυθεί τα κατάλληλα βήματα για να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και πληροφόρηση μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου και πρέπει η συνεργασία αυτή να ενταθεί ακόμη περισσότερο. Η διαφάνεια τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, όπω αναγνωρίζεται από τη συμφωνία, απαιτεί περαιτέρω προσπάθειε στη φάση υλοποίηση. Πραγματικά στα χέρια μας είναι να υλοποιηθεί αυτή η θεσμική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία με τρόπο ώστε να υπάρξει πολλαπλή προστιθέμενη αξία από αυτές τις προσπάθειες για να έχουμε καλύτερους νόμους, καλύτερο σύστημα δικαίου. Ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη συμμετοχή ε, τους, όλους τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα happy end σε όλη αυτή την προσπάθεια. Όπως είπατε πρόεδρε, είναι μόλις η αρχή μια υπέροχη κοινή προσπάθεια για την υλοποίηση αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Χιούμπνερ. Πιστεύω ότι όπως είπατε και εσείς πρόκειται για την αρχή μιας υπέροχης φιλίας. Μια φράση που γνωρίζουμε όλοι από την ταινία Casablanca, The Beginning of a Beautiful